Good morning, ladies and gentlemen. As we have very busy Έχουμε πάρα πολλή δουλειά σήμερα και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας, λέει Θα ξεκινήσουμε με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε κάποια σχόλια. Γίνεται δεκτή. Έγκριση των πρακτικών. 3 Δεκεμβρίου. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά online. Αν δεν ε, εκφραστούν κάποιες αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν ε, δεκτά. Τώρα οι ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν θα καθυστερήσουμε. Για το σημείο 4, την έκθεση την οποία πρέπει να ετοιμάσουμε για το πρόγραμμα συνεργασίας εδαφικής εδαφικής 4 Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας, Βορείου Ιρλανδίας, Σκοτίας, στα πλαίσια του θέματος της πιθανής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υπάρχει πρόβλεψη συνεργασίας και συνέχιση στον τομέα της διαμεθοριακής συνεργασίας. Δεν είναι σαφές όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επικυρώσει την συμφωνία αποχώρησης. Αν δεν υπάρξει τέτοια επικύρωση, αυτό θα δημιουργήσει θέματα στις μεθοριακές περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας που είναι συνέπεια και αποτέλεσμα της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής που οδήγησε στην ειρήνευση της περιοχής. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία πρόταση που προβλέπει μία απόκληση εξαίρεση έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα PIS4 στα πλαίσια των υπολείπων προγραμμάτων συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και ε, η Ιρλανδία στα πλαίσια της προγραμματικής περίοδου η οποία εξελίσσεται μέχρι δηλαδή και το 2020. Υπάρχουν άλλα 13 στα οποία συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αφορούν στην Ιρλανδία, οπότε δεν θα τύχουν της ίδιας εξαίρεσης. Η πρόταση συνεπώς προβλέπει την χρηματοδότηση του προγράμματος για τη Βόρεια Ιρλανδία στα πλαίσια του κανονισμού Interreg ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει ότι ε, δεν θα πρέπει άνω του προϋπολογισμού του 20% να δαπανάται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα εφαρμοστεί μιας ε, και η δαπάνηση κάποιων πιστώσεων στη Βόρεια Ιρλανδία θα ε, έπρεπε να περιοριστεί δραστικά. Λοιπόν δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας και είναι σαφές ότι ο κανονισμός θα πρέπει να υιοθετηθεί 4 πριν τις 30 Μαρτίου. Η Επιτροπή μας έστειλε μια αντιπροσωπεία στη Βόρεια Ιρλανδία το Μάρτιο του 2018 και στη συνέχεια ε, υπήρξε μια εφαρμοστική έκθεση του κυρίου Βόλτ ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι τα προγράμματα τα ειρηνευτικά θα πρέπει να διατηρηθούν και μετά τον Brexit ανεξαρτήτως του πλαισίου στο οποίο θα γίνει. Υπό το φως λοιπόν των αποφάσεων που πήραν οι συντονιστές την προηγούμενη εβδομάδα και ως εισηγήτρια σας προτείνω οι κανονισμοί αυτοί να, να αντιμετωπιστούν συγγνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 με την απλοποιημένη διαδικασία άνευ τροπολογιών. Η πρόταση εκθέσεως έχει ήδη διανεμηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους σας. Πριν προτείνω την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού, δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Βόλβε έχει το λόγο. Σύντομα, να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Όπως είπατε, εμείς ξεκινήσαμε με μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με την, την χρηματοδότηση των προγραμμάτων στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από το 2020, γι' αυτό έγινε και η αποστολή αυτή, η διερευνητική. Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής είδαμε πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα τα οποία διατηρούνται εν ζωή μέσω αυτής της χρηματοδότησης και όλα αυτά φυσικά αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στη Βόρεια Ιρλανδία την προηγούμενη εβδομάδα, ιδιαίτερα με τα τεκτενόμενα στην πόλη του Ντέρι. Ε, είδαμε πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση, μας είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό και το διαπιστώσαμε ήδη η σώμαση την εβδομάδα που πέρασε. Συνεπώς πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και μετά το 2020 Φυσικά είναι σημαντικό να πάει μέχρι το 20, αλλά πρέπει να παραταθεί. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Στο ίδιο πνεύμα και εγώ, όπως και οι προλαλήσαντες, κάναμε μία αποστολή εκεί και κάθε φορά γνωρίζαμε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαμε ε, έτσι και αλλιώς ε, πει ότι θα παρατείνουμε τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών. Διαπιστώσαμε ότι είναι εύθραστες οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και σε τοπικό επίπεδο και σαν παράδειγμα γίνονται προσπάθειες πάρα πολύ σημαντικές ακόμα και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού, προγράμματα συνεργασίας και γυτνίασης των δύο διαφορετικών πλευρών. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα αυτά Προγράμματα τα οποία έχουν προχωρήσει αρκετά βρίσκονται ορισμένα από αυτά στην τέταρτη φάση λειτουργία τους. Και ακούμε κάτι περίεργα πράγματα από το Λονδίνο σχετικά και με πιθανές αλλαγές στις προβλέψεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτά όλα θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν θέλουμε να τα φανταστούμε. Είναι απαραίτητο συνεπώς να υπάρξει αποδοχή ταχύτατη της πρότασής σας. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα PIS, αλλά ξέρουμε ότι αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα και το Ίντερνετ και ξέρουμε πώς το ντερεγ βοηθάει τα σχολεία ανάμεσα στις δύο μεθοριακές περιοχές α βοηθάει τις υποδομές, βοηθάει τις μεταφορές, γενικά την ανάπτυξη και των δύο πλευρών των σύνορων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν γιατί είναι και περιοχές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες. Υποστηρίζουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά την πρότασή σας λέει ο κ. Βανέστερόι. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοφτης έχει το λόγο. ως μέλος της αντιπροσωπείας που επισκέφτηκε τη Βόρεια Ιρλανδία. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Και έχουμε ακούσει και τις απειλές οι οποίες έχουν εξτομιστεί σχετικά με πιθανή πάυση της ισχύω ε, των συμφωνιών της Μεγάλης Παρασκευής. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή η οποία και αυτή είχε ε, προβλήματα διαχωρισμού, τείχους ε, και εμφύλια σύραξης, αιματηρής και δεν θα ήθελα να δω κάτι αντίστοιχο και στην Δυτική Ευρώπη. Εγώ έχω βιώσει την, τον εύθραυστο χαρακτήρα των σχέσεων στη Βόρεια Ιρλανδία φυσικά αλλά ξέρω πολύ καλά ότι οι νεότερες γενιές, ε, οι Ιρλανδοί και από τις δύο πλευρές θέλουν να ζήσουν σε, με ειρήνη και να αναπτυχθούν από κοινού. Λοιπόν, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, γιατί μία από τις δύο συμβαλόμενες χώρες στη συμφωνία αυτή ε, θα γίνει τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα. Είναι σημαντικότατη η περίοδος αυτή για τη συγκεκριμένη περιοχή και θέλω να υποστηρίξω τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υποστηρίξουμε όλους ε, στην Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία που επιθυμούν την ειρήνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή πράγματι είναι πολύ θετική, λέει ο κ. Χάουαρθ, και θα την υποστηρίξω. Είναι πολύ δύσκολη η εποχή για τη Βόρεια Ιρλανδία, για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας και για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πολλές από τις ε, απόψεις οι οποίες διαβάζεται... Ε, στην, ε, ε, στον τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου ακούγονται αστείες και ανεύθυνες. Πράγματι οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιαδήποτε πολιτικό κόμμα να σκέφτεται ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε μονομερείς αλλαγές στην συμφωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο καταδικάζω πλήρως και θα το καταδικάσουν και όλοι οι συνάδελφοί μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο μονομερός και όποιος ε, δίδει συμβουλές ε, στο γραφείο τύπου ε, του αριθμού 10 όπως λέγεται του Πρωθυπουργικού Γραφείου είναι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και μας εκθέτει σε κίνδυνο. Λοιπόν, ελπίζω η πρότασή σας να περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Ελπίζω να μην είναι κάτι το οποίο απαραίτητα θα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά σήμερα διάβασα άρθρα σχετικά με τις πιθανές οικονομικές ζημίες στις μεθοριακές περιοχές γύρω ε, από το θέμα της αποχώρησης. Μία από τις χώρες η οποία θα έχει πάρα πολλές ζημίες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι φυσικά η Ιρλανδία, όσο και αν οι Άγγλοι πολλές φορές αυτό δεν το συνειδητοποιούν. Συνεπώς λοιπόν η ειρηνευτική αυτή διαδικασία θα συνεχίσει ε, την ε, ειρηνευτική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ λέει κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για αυτά τα οποία είπαν. Εγώ είμαι από τον Τέρι, λέει η κυρία Άντερσον. Ε, είμαι από την περιοχή από την οποία προέρχεται και ο Μάτι Μαγκίνες. Ε, είναι η πόλη στην οποία εξεράγει μια βόμβα την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ε, χτες είχαμε επίσης κάποιες απαγωγές στον Τέρι, κάτι το οποίο δεν είχαμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είχα απαχθεί στο παρελθόν, είχα κρατηθεί παρανόμως στις φυλακές και από τότε που απελευθερώθηκα από τη φυλακή έκανα καθημε, κάνω καθημερινές προσπάθειες για την προστασία της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η απαράδεκτη καταδικαστέα συμπεριφορά της Βρετανικής κυβέρνησης είναι έτοιμη να την άξει στον αέρα το Ηνωμένο Βασίλειο και να παραβιάσει τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι σκανδαλώδες αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες, βάσιμες ανησυχίες και ήρθατε στον Τέρι, είδατε την κατάσταση, πήγατε στον Μπέλφαστα, συναντηθήκατε με τους υπευθύνου και είδατε την εξαιρετική δουλειά την οποία προσφέρει στην περιοχή το πρόγραμμα Interreg σαν παράδειγμα είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία βοηθά την ειρήνευση και τη συμφιλίωση η οποία προχωρά σταθερά αλλά με χαμηλές ταχύτητες και θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή και γνωρίζω και αυτά τα οποία είπατε για τα υπόλοιπα 13 προγράμματα και στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου και στα πλαίσια του Περιφερειακού Ταμείου τα οποία τα χρειάζεται η περιοχή έτσι ώστε οι δύο πληθυσμοί να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Θα συζητήσουμε αναλυτικότερα τις επόμενες μέρες την οικονομική ζημία την οποία θα έχει προκαλέσει η πιθανή αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η Βρετανική κυβέρνηση να αγνοήσει και να παραβιάσει την ε, συμφωνία της Μεγάλης ε, Παρασκευής. Και έτσι και αλλιώς βέβαια εξαρτάται μένα από το Democratic Union Party, το DUP, η επιβίωση της κυβέρνησης της κυρίας Μέη, αλλά να θυμίσουμε ότι το DUP σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρ και δεν υποστήριξε ουσιαστικά τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να μην ε, διακόψουμε τις ε, συνθήκες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο περιοχές της Ιρλανδίας και ακριβώς η Μεγάλη Παρασκευή, η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής έχει επιτρέψει την απρόσκοπτη επικοινωνία. Δεν θέλω να υπερδραματοποιήσω τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει τα διάφορα τμήματα της Συμφωνίας ε, της Μεγάλης Παρασκευής και να μην υποστηρίζει αυτά τα οποία επιθυμεί σε σχέση με τη συμφωνία αυτή ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας είναι αγανακτισμένος με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει λοιπόν ε, ε, είναι σαφής ε, η επιθυμία των λαών της περιοχής, η δημοκρατική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ε, τις διαδικασίες αυτές από τον προηγούμενο Απρίλιο. Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας και την καταδικάζω, αλλά οι δημοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει παρακαλώ να συνεχίσετε να επιτρέπετε στους λαούς της Ιρλανδίας να συνεχίσουν τις επικοινωνίες μεταξύ τους και αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποια ένωση θέλουν να συμμετέχουν από τις δύο που προσφέρονται και θέλουν φυσικά να διατηρηθεί η σχέση που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Λοιπόν δεν άκουσα καμία αντίρρηση για την πρόταση την οποία έκανε σχετικά με την έκθεση αυτή. Συνεπώς η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, για να υπάρξει μια απόκληση εξαίρεση ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέχρι το 2020 μπορεί να θεωρηθεί δεκτή. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα εδαφικά προγράμματα συνεργασίας στη Βόρεια Ιρλανδία στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής την οποία μόλις λάβαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεκτή η ε, πρόταση εκθέσεως τώρα. Περνάμε στις ψηφοφορίες. γνωμοδότησε της Επιτροπής Ρέτσι για την διαδικασία απαλλαγής για το 2017 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συναρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Κόντ και ως ε, συντάκτρια συζητήσαμε την γραμμή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 Ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση για το νέο κανονισμό περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021 με 2027. Όπως γνωρίζετε είναι, ένα, μία από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, πολιτική σύμβουλοι, εισηγητής, συνεισογητές, ε, στελέχη της γραμματείας. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν δουλέψει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες για να ε, οργανώσουν αυτή την ψηφοφορία. Έχουμε πάνω από 2.000 τροπολογίες και τις τροπολογίες των 10 ε, συναρμοδίων επιτροπών που έχουν συντάξει γνωμοδοτήσεις. Είναι μια ψηφοφορία η οποία θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προτείνω λοιπόν ε, περίπου στη μέση να κάνουμε διάλειμμα λίγων λεπτών. Θα σας πω πότε για να δούμε και πώς θα έχει προχωρήσει η ψηφοφορία μέχρι τότε. Άρα, όλο το σημερινό πρωινό θα το αφιερώσουμε σε αυτή την ψηφοφορία. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, δίνω το λόγο στους συνεισηγητές. Η κυρία Κρέλου, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω ήδη ακούσαμε, κατατέθηκαν πάρα πολλέ τροπολογίε. Έχουμε τι γνωμοδοτήσει πολλών διαφορετικών επιτροπών. Τι επεξεργαστήκαμε και πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντατική, αλλά και πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους σκιώδους συζητητές. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όχι μόνο τους ε, σκιώδους συζητητές, αλλά και την Γραμματεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλες τις πολιτικές ομάδες, τους βοηθούς, τους υπαλλήλου, χωρίς την υποστήριξη των οποίων ε, και χωρί όλε αυτέ τι ώρε που κάτσαν και δούλεψαν, δεν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Σκοπό μα, σκοπό των δύο συνεισηγητών, είναι σε υψηλό επίπεδο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Όσο πιο καλή ποιότητα διαπραγματεύσει γίνεται. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα ωφελήσει, θα ωφελήσει και τις ε, περιφέρειες. Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι είναι έτοιμο να συζητήσει τους τριμερείς διαλόγους μαζί μα για τα θέματα του προγραμματισμού και πιστεύω ότι είναι δικό μα ε, καθήκον να ξεκινήσουμε αυτού του ε, δύο τομεί και να του ολοκληρώσουμε αυτού του δύο τομεί όσο πιο γρήγορα γίνεται για να δώσουμε την ευκαιρία στι περιφερειέ να ξεκινήσουν και να καταστρώσουν τα δικά του ε, λειτουργικά προγράμματα και να υπάρξει αυτή η αναδιάτρωση. Γι' αυτό λοιπόν θερμοπαρακαλώ, παρακαλώ τους συναδέλφους. Πετύχαμε πάνω από 100 συμβιβαστικέ προτάσει. Συμβιβαστικέ προτάσει που όπω το λέει και η λέξη δεν θα του ικανοποιήσουν όλου κατά 100%. Δεν ε, ε, περιλαμβάνεται καν αυτό που ήθελα εγώ κατά 100% σε αυτή την πρόταση. Αλλά στο τελική ανάλυση αποτελεί ένα συμβιβασμό. Και το Κοινοβούλιο κατεξοχήν ε, έχει αναπτύξει μία κουλτούρα προσέγγισης αλλήλων. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλώ τους συναδέλφους ακόμα και αν δεν είσαστε 100% ικανοποιημένοι να υπερψηφίσετε τελικά την έκθεση αυτή προκειμένου με συντριπτική πλειοψηφία να πάμε στην Ολομέλεια και να πούμε ότι κοιτάξτε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξη υποστηρίζει στεναρά αυτή την έκθεση. Αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή καθόλου δεδομένο. Για να ξεκινήσουν λοιπόν και οι διαπραγματεύσει μετά την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Αυτό θα σα παρακαλούσα και αν έχετε οποιαδήποτε τελευταίο δισταγμό να τον υπερπηδήσετε γιατί η δουλειά που κάναμε από κοινού είναι σημαντική. Και να ψηφίσετε αντίστοιχα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Και εγώ ευχαριστώ, κύριος Νοβάκοφ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο Λίγοι από εσά νόμιζαν ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε στην Ολομέλεια ένα τέτοιο και κείμενο. Χαίρομαι γιατί πολλοί από εσά αλλάξατε γνώμη και στηρίξατε τι προσπάθειέ μα. Κάναμε όλοι πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο τη ψηφοφορία στην Επιτροπή μα. Είναι μια ιστορική ευκαιρία να κάνουμε ένα άλμα προ τα εμπρό, να ψηφιστεί στην Ολομέλεια και να ξεκινήσουμε την επαύριο διαπραγματεύσει αμέσω. Και η Ρουμανική Προεδρία έχει διακηρύξει την ετοιμότητά τη ω προ αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα, να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις των διαφόρων δικαιούχων απανταχού στην Ευρώπη και πρέπει να εγγυηθούμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε η επόμενη προγραμματική περίοδος να ξεκινήσει ομαλά 1η Ιανουαρίου του 2021. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και για να το καταφέρουμε ζητώ τη στήριξή σας να ψηφίσετε τις συμβαστικές τροπολογίες και τελικά την, ε, το σύνολο του κειμένου και να το υπερψηφίσετε και στην Ολομέλεια, την επόμενη Ολομέλεια. Θα είναι το δικό μας κοινό επίτευγμα, η δική μας κοινή τύχη, ο δικός μας επιτυχημένος αγώνας με αντίπαλο το χρόνο χρειάστηκαν πάρα πολλές προσπάθειες και πολύ μεγάλη και πολλή δουλειά έτσι ώστε να συγκεραστούν όλες οι απόψεις και να φτάσουμε σε ένα σταθμισμένο ε, τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης έτσι ώστε όλοι ε, να βλέπουν στο κείμενο ότι οι ανησυχίες τους και τα αιτήματά τους και οι ανάγκες τους έχουν καλυφθεί και πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα νησιά, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, περισσότερο ανεπτυγμένε περιοχές. Όλα τα συμφέροντα όλων των πολιτών ε, αντικατοπτρίζονται και απεικονίζονται στην έκθεση αυτή. Ελπίζουμε να έχουμε τελικά την πλειοψηφία και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το κείμενο στην Ολομέλεια. Ένα θερμό ευχαριστώ στου συνεισηγητέ, στου κοιόδη εισηγητές και στη συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω. Ελέγχοντας τις παρουσίες ε, στην αίθουσα των συνεδριάσεων και συσκέψεων, να σας πω ότι ίσως έχουμε μόνο δύο ψήφους από την ομάδα των Πρασίνων και το ξέρετε εσείς αυτό. Καλώς. Το λέω γιατί είστε τρεις εδώ. Ευχαριστώ. Πρέπει συνεχώς να μετράω και να υπολογίζω. Ε, νομίζω ότι στηρίζετε πολύ την έκθεση και εσείς η ομάδα σας είναι εδώ. Καλώς. Ξεκινούμε λοιπόν την ψηφοφορία. Έγκαιρα, ακριβώς όπως είχαμε ξεκινήσει, στις 9, όπως είχαμε προγραμματίσει στις 9 και μισή. Συμβιβαστική Α1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική, στην α2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 6 συν 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Που είναι κάπου πιο μετά. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 συν 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Συμβιβαστική 7 θα είναι η επόμενη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Προχωράμε, προχωράμε στην 9 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α11 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική α12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία έκον 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 749 υπέρ, κατά. Άποχες Απορρίπτεται. Στη ΛΥΜΠΕ 52 πάμε. Όχι. Ναι. Η Α14 καταπίπτει. Α14, ναι, καταπίπτει. Άρα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται η Α14. Α15 συμβαστική, ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε το επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε την Α15 ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ 15 κατά. Συμβιβαστική Α16. Λίγο πιο πέρα είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 974. 974 για να τη βρω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 974 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Συμβιβαστική Α18. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 παύλα 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 κάθετος 2 καταπίπτει. Και πάμε τώρα στην 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα του καταλόγου ψηφοφορίας. Πολύ καλή δουλειά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Τα επαναλαμβάνω όλα αυτά γιατί έχετε λάβει τους καταλόγους ψηφοφοριών ανατμήματα και γι' αυτό αναφέρω τα τμήματα, να ξέρετε ποιο ε, φυλάδιο βγάζετε. Α22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α23 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α α25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 16 της ένβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12.96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.97 και 81 της Λίμπε. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12, 96 και 75 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνονται. Της η 82 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 1338 της ΦΕΜ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 83 της ΛΥΜΠΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Α37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 22 της ΛΥΜΠΕ, 86, 1332 και 41 της ΦΕΜ, της Επιτροπής Γυναικών. Όλες αυτές μαζί. Και, όχι είναι άλλη αυτή. Αυτές οι τέσσερις που είπα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Πάμε τώρα στην 1323. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13, 24 και 40 της ΦΑΜ. Μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 87 της ΛΥΜΕ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13-25 υπέρ, κατά, αποχές απορριπτεται 13.26. υπέρ. Κατά. Αποχές. 13.28. υπέρ. Κατά. Αποχές. 13.30 και 88 της Λίμπε. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1331 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 33 καταπίπτει. 1334 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1336 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1337 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1338 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 91 της Λίμπε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1369 μαζί με 1371 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 1370 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εκρίνεται, αλλά στο το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. 13.70. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία εβδομήντα δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 αποσύρεται 1373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1378 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13.79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13.80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 13 91 λέει η συγγήτρια. Υπέρ η πρόεδρος. Κατά αποχές απορρίπτεται. Α52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α54 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1393 κάθετος 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1424, υπέρ. Κατά. Αποχές 1426. υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτεται 1425. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1423. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσύρεται η 27, πάμε στη 14-28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14-30. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14-31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1435 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην τραν 35 λέει η συγκήτρια υπέρ κατά Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Τραν 35. Υπέρ. Κατά. Τραν 35. Λοιπόν, έγινε μπέρδεμα να δούμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την Τραν 35. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Καλώς, ευχαριστώ. Συμβιβαστική Α58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1449 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 1449. Καλώς. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 14.50. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1452. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 1453. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1454 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 1454 απορρίφθηκε. Καταπίπτει λοιπόν τώρα, γι' αυτό πάμε στις τρεις τροπολογίες 1455, 1464 και 1463. Ποιος είναι υπέρ, τη ψηφίζουμε μαζί. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική α62 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. α63 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 5007. 15.07. 15.07. Λόγω των προηγουμένων ψηφοφοριών ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Στη 15.07 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική α64. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15.08. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1509. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1510. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 της Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ταυτόσημες η 11 η 45 της ΦΕΜ, η 12 και η 107 της ΛΥΜΠΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 15-13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15-14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 15-15. Υπέρ. αποχές ε, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν από εκείνο το 15-16 και την άγκρη 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 15-18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15-19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Α67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1571. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Α70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15.82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15.83 και λίπε 110. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15.84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 34 της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1586. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1587. 1587 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1590 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1591 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1592 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1593 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 15.95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 15.96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15.97. Και λίμπε 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 1599 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1601 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1602 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16-17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16-18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική α84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α85. Πολλές σελίδες. Πολύ ωραία. Προχωράμε. α85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. α86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96 μαζί με την 1759. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1760. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1761. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1762. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική α90, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α91, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1774. Αποκινούμε τη λίμπα 115. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17.75 και 17.76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17.78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17.79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε από κοινού. τεσσερι τροπολογίε. 17, 1781, 1782, 1783. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική Α99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18-10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α104 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική Α105. Και πάλι περνάμε πολλές σελίδες. Α105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α106. Κάθετος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην α106 κάθετος 2. Υπέρ. Η α106 κάθετος 2 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε έναν έλεγχο για την α106 κάθετος 2 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ξέρετε τι ψήφισε ο καθένα. Μάλιστα. Αν όλοι ξέρετε τι ψηφίσατε. Πολύ εντυπωσιακό. Τι να πω. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η συμβιβαστική και άρα συνεχίζουμε με το 16-20. Τροπολογία 16-20. Μια και απορρίφθηκε ο συμβιβασμό, συνεχίζουμε και ψηφίζουμε τι επιμέρου τροπολογίε. 16-20 λοιπόν υπέρ. Να σας εξηγήσω, λέει η Πρόεδρος. Εφόσον απορρίψαμε τη συμβαστική πρόταση, την υπαριθμόν 106 ε, 2, καλούμαστε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες που καλύπτονταν προηγουμένως από τη συμβαστική πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε την 16-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι άλλε δύο καταπίπτουν λόγω τη προηγούμενης ψηφοφορία Η 120 λοιπόν, η επόμενη. Καταπίπτει επίση. 121. Ψηφίζουμε την ε, Άγκρη 41 τώρα. Άγκρη 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2004. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20.05 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές και νομίζω ότι καταπιπτεί. Μάλλον απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο τρίτο τμήμα. Μήπως θέλετε να κάνουμε διάλειμμα.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 η τροπολογία της Λίπε για τον άρθρο 13. Άρθρο 13 παρακαλώ, για ψάξτε στην παράγραφο 2. Πολύ λυπάμαι γιατί δεν έχουμε αριθμό σελίδων. Αυτό γιατί έγιναν και τελευταίες αλλαγές. Άρθρο 13 παράγραφος 2. Το βρήκατε παρακαλώ. 13, παραγραφός 2. Έχουμε δύο τροπολογίες. Απορρίψαμε την πρώτη, την, 10, την 749 και γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε τη Λίμπε 52. Αν τη βρήκατε παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ για τη ΛΥΜΠΕ 52. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι με τα δύο πρώτα Αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι, δεν θέλετε. Πολύ ωραία. Πάμε στα παρατήματα. Αιτελογικές σκέψεις. Και γι' αυτό λοιπόν έχει διαφορετική αρρύθμιση πλέον ε, η κάθε συμβαστική πρόταση. Χ1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 88 της Επιτροπής Απασχόλησης. Τώρα. Τροπολογία 88 της Επιτροπής Απασχόλησης. Με την 80, 90, 91 και 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 21-43 υπέρ. Κατά. Αποχές και νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για το 21-43? Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Και σας ευχαριστώ. 21-43 λοιπόν εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην 125 και την 20.07. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 20.07, Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 2009 υπέρ. Κατά. Αποχές 21 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2012 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 2148 μαζί με την ΦΕΜΑ 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η 2150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 21 2149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 Καταπίπτει. Employment 94. Υπέρ. Υπέρ για την 94 της Επιτροπής Απασχόλησης. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 94 ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την 2152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2155. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 2157. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος στείτε για την 2159. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. περασε Εγκρίνεται. 21.60. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 21.61. Από κοινού με την 366. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21.62. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 21-63. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τραν. 67. κάθετο 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τραν 67. κάθετο 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τραν 67 κάθετος 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 64 κάθετος 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τραν 67 κάθετος 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τραν 67 κάθετος 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τραν 67 κάθετος 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2164 κάθετος 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τραν 67 κάθετος 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τραν 67 κάθετος 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21.65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 21.66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 21.67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21.68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2170 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2170 ψηφίζεται τέλος της ψηφοφορίας δεκτή 2169 υπέρ κατά αποχές δεκτή. έμπλε 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή. έμπλε 96 υπέρ κατά αποχές δεκτή. έμπλε 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. έμπλε 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έμπελε 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2171 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2172 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2173 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2174 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2175 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 2175 ψηφίζεται Πέρας της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή. Έμπλ 100. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2176. Υπέρ. Κατά. αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2177 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2178 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21, 80 και 81 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 2179 και έμπλε 105 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Έμπλε 108 και 109 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2013 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2014 και 2015 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή μαζί οι 128 και οι 2016 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτε, απερίφθησαν. ΕΜΠΛΕ 111 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 129 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2017 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Λίμπε 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απερίφθη, απερίφθη λέει η προεδρο συγγνωμη συγγνώμη, απερίφθη. 20-19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 20-20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 20-21 υπέρ κατά, αποχές, απερίφθη. έξι ταυτόσομες, η 1, η 132, η 133, η 134, η budget 1, η agri 1, Ένα, συγγνώμη, υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Τώρα η λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική R αγγλικό 1 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική R1 α κεφαλαίο υπέρ κατά αποχές, δεκτό. Συμβιβαστική R2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λίμπε 7, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική R4, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική R5, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 167 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική R9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική R10 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική R11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 200, 201, 202 και 203 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική R13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. R14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στη συμβιβαστική R20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική R20 α κεφαλαίο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λίμπε 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Συμβιβαστική R23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 277 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 277. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική R27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 282 μαζί με την ΦΕΜ 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΕΜΠΛ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική R30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΛΥΜΠΕ 21. Υπέρ κατά, αποχές, απερίφη. Συμβιβαστική R34 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστη... μάλλον η 286 μαζί με την κοντ 4 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική R36 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική R38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 291 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική R40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 296 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 2.97 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.98 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων. Είναι κάποιος κατά? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λίμπε 25 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Ψηφίζουμε από κοινού λοιπόν την 301, τη ΛΥΜΠΕ 26, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Συμβιβαστική R46, υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 305, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική R48α κεφαλαίο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 310 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 311 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική R50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.13 αποκινούμε την κοντ 6 υπέρ κατά αποχές δεκτές συγγνώμη για μια στιγμή η 3-13 μαζί με την κοντ 6 απερίφθησαν συμβιβαστική R58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη απερίφθη υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική R61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 322 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική R63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 330 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Τροπολογία 331 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 331, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. Συμβιβαστική R66α κεφαλαίο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα περνάμε στην τελική ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες Η έκθεση γίνεται πλέον δεκτή. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους συμβούλους, τις πολιτικές ομάδες και όλους όλους εσάς για την προσπάθεια που κάνατε σήμερα. Εμείς ολοκληρώσαμε λοιπόν τις, ε, την ημερήσια διάταξή μας για, για το πρωί. Θα κλείσει τώρα η συνεδρίαση και θα συναντηθούμε στις 3 το μεσημέρι ε, με την Ρουμανική Προεδρία.